przewodniczący! Good morning, Καλημέρα, παρακαλώ να πάρετε τη θέση σας. Αρχίζει η συνεδρίασή μας. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τα συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 28-29 Οκτωβρίου και οικονομική διακυβέρνηση. Υποδέχομαι και χαιρετίζω την παρουσία στην αίθουσα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κ. Χέρμαν Βανομπόγιου και την παρουσία επίσης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Χωσέ Μανουέλ Μπαρόσο. Επίσης μεταξύ μας έχουμε τους εκπροσώπους της Βελγικής Προεδρίας και Επιτρόπους. Θα αρχίσει η συνεδρίασή μας με μία ενημέρωση και κατόπιν την ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κυρίου Βαν Ρομπόι. Περίμενε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28 και 29 Οκτωβρίου εστιάστηκε στην οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης ειδικότερα βάσει της έκθεσης της Ομάδας Εργασίας για την Οικονομική Διακυβέρνηση. Η έκθεση εγκρίθηκε. Και θα αναφερθώ ειδικότερα στην Ιρλανδία, τονίζει τη σημασία του θέματος γενικότερα και την ανάγκη για έναν μηχανισμό που να μπορεί να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί άμεσα. Χαιρετίζω την ταχύτατη αντίδραση των Υπουργών Οικονομικών και τονίζω ότι αυτό δείχνει το επίπεδο αποφασιστικότητας όλων των ενδιαφερομένων προκειμένου να διαφυλαχθεί η σταθερότητα του ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη θα δώσουν οικονομική υποστήριξη στα πλαίσια ενός ισχυρού προγράμματος πολιτικής που θα διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ιρλανδία, την, τον και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασιστική εφαρμογή αυτού του προγράμματο ελπίζουμε ότι θα επιτρέψει την επιστροφή σε σταθερή και στεναρή οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Αναφέρομαι στις πρωτοβουλίες τη Eurogroup και του ECOFIN. Δεν πρόκειται για διακυβερνητική διάσκεψη, αλλά για μια αναθεώρηση των μεθόδων εργασίας, των προτεραιοτήτων και των διαδικασιών μας αναζητήσαμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε ένα ευρύ ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα καταπολεμούσε τις ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ θα επιτρέπει σε εθνικές κυβερνήσεις ελεύθερα να αποφασίζουν τι θέλουν να δαπανίσουν σύμφωνα με τις εθνικές τους πολιτικές διαδικασίες. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε κράτος μέλος θα λαμβάνει απόλυτα υπόψη τις επιπτώσεις των οικονομικών και δημοσιονομικών αποφάσεων για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Ταυτόχρονα θέλουμε να ενισχύσουμε την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδρά όταν οι πολιτικές σε ένα κράτο μέλος αποτελούν, σημαίνουν κίνδυνο για τα υπόλοιπα κράτη μάλλη. Οι συστάσεις της ομάδας εργασίας είναι πολύ κοντά στις προτάσεις της Επιτροπής. Συζητήσαμε τα θέματα αυτά δύο φορές με τους επικεφαλείς των ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τους προέδρους των αρμοδίων επιτροπών. Ε, ε ανταποκρινόμενοι στο αίτημά σας. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι απογοητεύθηκαν, διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος αυτοματισμός στη διαδικασία λιάψοφάσεων. Περισσότερος αυτοματισμός είναι ακριβώς αυτό που προτείνουμε. Το Συμβούλιο, το Συμβούλιο βάσει της συνθήκης αποφασίζει για κυρώσεις βάσει μιας όπως ονομάζεται δυσοφής πλειοψηφίας. Δηλαδή αν δεν υπάρχει δική πλειοψηφία κατά ε, θα ισχύσουν οι κυρώσεις ενώ τώρα η πλειοψηφία έπρεπε να τις εγκρίνει. Πριν από λίγες εβδομάδες μόλι ορισμένα κράτη-μέλη δίσταζαν για αυτή την ε, αντίστροφη ε, πλειοψηφία και η ομάδα εργασία πρότεινε μια σειρά από άλλα μέτρα που έχουν σκοπό να ενισχύσουν το σύμφωνο σταθερότητα. Περισσότερο συντονισμό των πολιτικών, το ευρωπαϊκό εξάμεινο, υγιεί ε, στατιστικέ και δημοσιονομική έλεγχη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι οι αποφάσει που λαμβάνουν επηρεάζουν όλα τα κράτη-μέλη τη Ένωση. Αυτό είναι το σημαντικό δίδαγμα που πήραμε από την κρίση. Η ομάδα εργασίας ήταν ένα πολιτικό πλαίσιο που είχε σκοπό να εξασφαλίσει γρήγορη συνένεση. Όλες οι πρόοδοι που σημειώθηκαν πρέπει τώρα να μεταφραστούν σε νομοθετικά κείμενα. Η δουλειά αυτή θα γίνει από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Όλα τα θεσμικά όργανα θα διατηρήσουν την αναγκαία όθηση και θα αναλάβουν πλήρω τι ευθύνε του. Το κύριο στοιχείο τη ομάδα εργασία και είναι σημαντικό για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θέλουμε έναν στεναρό μηχανισμό ε, διαχείριση κρίσης για να διαφυλαχθεί η σταθερότητα τη Ευρωζώνη και τη Ευρώπη γενικότερα. Όλα τα αρχηγοί κρατών συμφώνησαν γι' αυτό πριν, προτού ολοκληρώσουμε γι' αυτό το σημείο, θέλω να υπογραμμίσω ότι η δουλειά για το σύμφωνο σταθερότητας δεν αφορά την επιβολή κυρώσεων στα κράτη-μέλη ή τη διόρθωση των λαθών του παρελθόντος. Πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη σημαντική πρόκληση για τη βελτίωση της σταθερής ανάπτυξης της Ευρώπης και των γενικών οικονομικών επιδόσεών της. Σε αυτό εστιάστηκε η στρατηγική του 2020 που ενέκνεσε στις αρχές αυτού του έτους το Συμβούλιο. Η απάντηση εκείνων που φοβούνται ότι η δημοσιονομική λιτότητα θα εμποδίσει την ανάπτυξη και θα επηρεάσει τους διαφορετικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις οικονομικές επιδόσεις μας θα είναι ο κύριος στόχος των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου του χρόνου. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε επίση μια σύντομη συζήτηση για τα θέματα του ευρωπαϊκού προπολογισμού μετά από την ομιλία του Προέδρου σας στην έναρξη της συνεδρίασής μας. Στο μεταξύ τα συμπεράσματά μας λένε ότι είναι σημαντικό το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δημοσιονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο να υπογραμμίζουν τις προόδους που έχουν σημειώσει τα κράτη-μέλη για να περιορίσουν το έλλειμμα και το χρέος σε πιο λογικά επίπεδα. Υπογραμμίζω, σεβόμενοι το ρόλο των διαφόρων θεσμικών οργάνων και την ανάγκη να ανταποκριθούν στου στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο θα συζητήσει στην επόμενη συνεδρίασή του πώ θα εξασφαλιστεί ότι οι δαπάνε σε ευρωπαϊκό έπεδο μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα να σα διαβεβαιώσω και πάλι ότι αναγνωρίζουμε τον νέο ρόλο του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Βεβαίω δεν πήραμε θέση ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον προπολογισμό του 2011. Αυτή είναι μια διαδικασία που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Πάντως, απευθύνομαι σε όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τους προκειμένου να επιτευχθεί μια συμβιβαστική λύση για τον προπολογισμό του 2011 το ταχύτερο δυνατό στο συμβιβασμό όλα τα, όλες, όλα τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να ληφθούν υπόψη ενώ θα τηρείται και θα γίνεται σεβαστή στην θήκη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως συμβαίνει και με όλα τα ευρωπαϊκά συμβούλια, επέτρεψε την επίτευξη κοινών θέσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση για σημαντικά διεθνή θέματα. Η προσοχή μας εστιάστηκε στην προετοιμασία της συνάντησης του G20, την ε, διάσκεψη για το κλίμα ε, της Κανκούν και για σε άλλα θέματα για την, σε ό,τι αφορά το G20 συμφωνήσαμε για τις προτεραιότητες που προωθήθηκαν στου προσώπους της Ένωσης και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στη, στο G20. Έγκριση το, του θέματος τη, το, της κεφαλαϊκής απάρκειας και της Προεδρίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτά κατέστησαν δύνατα λόγω της επικοδομητικής στάσης που τήρησαν οι Ευρωπαίοι. Παραχωρήσαμε δύο θέσεις για να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία στα πλαίσια της ε, προσπάθειας προσαρμογής. Σε ό,τι αφορά τις ανισότητες, την πολιτική των ε, ε, συναλλαγματικής πολιτικής κλπ. Η Σύνοδος Κορυφής κατέληξε σε μια διαδικασία μετά από εμπεριστατωμένη ανάλυση θα έχουμε μία σειρά από δείκτες για τις ανισότητες που θα προωθηθούν το 2011. Τώρα είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα και σε διορθωτικά μέτρα με βάση αυτή την αξιολόγηση. Για το Κανκούν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προετοίμασε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν στο τέλος αυτού του μήνα. Μετά την Κοπενχάγη πέρσι, Πάρα πολλέ συνομιλίε έχουν λάβει σε ε, χώρα σε άτυπο ή επίσημο επίπεδο. Οι απόψει διαφέρουν σημαντικά. Το Κανκούν θα είναι ένα ενδιάμεσο βήμα για ένα τελικό ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. θα συμβάλλει βεβαίως σε αυτή την προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διμερεί θέματα. Συζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Προτεραιότητας και Στρατηγικές για τις επερχόμενες συνόδους κορυφής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Ινδία και την Αφρική. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τον πρόεδρο Μπαρόσο και μένα και εξασφαλίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα μιλάμε όχι μόνο για τα θεσμικά όργανα των Βρυξελών αλλά και για τα 27 κράτη-μέλη συνολικά. Αυτό θα αποτελέσει τακτικό στοιχείο των μελλοντικών συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εδώ ολοκληρώνεται, αγαπητοί συνάδελφοι, οι συνάδελφοι τη τελευταία συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έλαβε χώρα πριν από περίπου ένα μήνα. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσω να εφαρμόζω την πρακτική μου ε, που είναι να ενημερώνω τους αρχηγούς των ομάδων ε, λίγη ώρα μετά τη λήξη κάθε συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και προσβλέπω στη, στο να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστούμε Πρόεδρε για την ομιλία σας. Τώρα θα ήθελα ο κύριος Πρόεδρος Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, εξότιμα μέλη. Όποιο είναι πολύ καιρό στον χώρο τη πολιτική βλέπει τι έχει συμβεί και πόσο σημαντικά είναι τα πρόσφατα γεγονότα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η δράση που έχουμε σχεδιάσει είναι ένα περαιτέρω αποφασιστικό βήμα για να εξασφαλίσουμε την οικονομική σταθερότητα τη Ιρλανδία, τη Ευρωζώνη και γενικότερα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δύο εργαλεία που θεσπίστηκαν τον Μάιο είναι αποτελεσματικά. Πραγματικά εργαλεία που θέλουν να φέρουν ει πέρα στο έργο που έχουν αναλάβει η Ιρλανδία. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και τα εργαλεία αυτά μπορούν να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Η παρέμβασή μα θα πρέπει να επιτρέψει στην Ιρλανδική οικονομία να ανακάμψει, να φτάσει στη τη βιώσιμη ανάπτυξη και να αναπτυχθεί, ανακτώντα την ζωτική τη δύναμη. Πρόεδρε, εξότιμα μέλη. Του περασμένου μήνε αντιμετωπίσαμε πολλέ προκλήσει. Κάναμε πολλή προσπάθεια, όμω για την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο μα. Η οικονομική διακυβέρνηση μεταρρυθμίζεται αυτή τη στιγμή ομάδα δράση όπου προεδρεύει ο πρόεδρο Φαν Ρόμποϊ έχει δώσει ήδη τα πρώτα, τους πρώτους καρπούς των έργων τη, που είναι πολύ αισιόδοξα. Ε, Βλέποντα λοιπόν και τη συνεισφορά τη Επιτροπή, βλέπουμε ότι έχουμε πετύχει μεγάλη σύγκληση στι ε, νομοθετικέ προτάσει τη Επιτροπή και έχουμε καλύψει και άλλου πολύ σημαντικού τομεί τη οικονομική διακυβέρνηση. Κατά κύριο λόγο, αυστηρότερου φορολογικού κανόνε και ευρύτερη οικονομική οικονομικό έλεγχο καθώς και το πακέτο των ε, θεσμικών μέτρων. Όλα αυτά διαφυλάχθησαν. Όπως τονίσαμε πολλές φορές στο παρελθόν, η σημασία το να έχουμε ένα πλαίσιο που να λειτουργεί άμεσα είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να στηρίξει την ιδέα μας για μια διαδικασία ταχείας προσέγγισης και να πετύχουμε του στόχου μα για συμφωνίε στι νομοθετικέ προτάσει τη Επιτροπή το, μέχρι το καλοκαίρι του 2011. Οι ερωτήσει που τέθηκαν και οι απορίε που τέθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο προ την ε, Επιτροπή και για το πότε θα υποβληθούν νομοθετικέ προτάσει από την δική μα πλευρά, τώρα έχουν μεταφερθεί και μεταφερθεί σε επιθυμία να περάσουμε στη διαδικασία αυτή τη ταχεία προσέγγιση. Για του προσεχεί μήνε Πρέπει να εργαστούμε αποτελεσματικά στο Κοινοβούλιο, όπω έχει γίνει ήδη στο παρελθόν, και να μα βοηθήσετε κι εσεί να στηρίξουμε την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω, είναι πεποίθησή μου, ότι θα καταλήξουμε σε σκληρού κανόνε που θα βασίζονται σε απαραίτητα κίνητρα για την συμμόρφωση, στην ε, ημιαυτόματη ε, εφαρμογή και ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ώστε να διορθωθούν ε, τα οικονομικέ διαφορέ ανισορροπίε. Πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση για να έχουμε βιώσιμη και αποτελεσματική πραγματική οικονομική ανάπτυξη, κάτι πολύ σημαντικό για το όφελο και το συμφέρον όλων των πολιτών μα. Ε, πρόεδρε, εξωτήμα μέλη. Ο μηχανισμός ε, για την Ευρωζώνη είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ε, λιθαράκι όλου αυτού του οικοδομήματος. <clears throat> το σύστημα που σήμερα ισχύει θα λήξει το 2014. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα αξιόπιστο ε, και εύρωστο σύστημα που να λειτουργεί ω τότε για να αντιμετωπίσει τις νέες οικονομικές πραγματικότητες. Η Επιτροπή ήδη έχει ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές τη εργασίες μελετώντα τα γενικά στοιχεία ενό μελλοντικού μηχανισμού για την Ευρωζώνη ο μηχανισμό αυτό, τον οποίο προετοιμάζουμε σε στενέ διαβουλεύσει με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα πρέπει να ε, γίνει αντιληπτό σε ένα μέρο του γενικότερου πλαισίου να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Θα ήθελα λοιπόν να καταστήσω σαφέ ότι ακόμη και αν ο μηχανισμό ε, χρηματοδοτηθεί από εθνικού προπολογισμού, θα παραμείνει μια βασική πρωτοβουλία ευρωπαϊκή που θα πρέπει να βασίζεται στην εμπρογνωμοσύνη, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία τη Επιτροπή, ώστε να μπορέσει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο μηχανισμό θα έχει τρει βασικέ συνιστώσει μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής, οικονομικούς διακανονισμούς και την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Το τελευταίο θα μπορεί να λάβει πολλές μορφές. Αλλά κατά κύριο λόγο θέλω να καταστήσω σαφές ότι ό,τι και αν αποφασιστεί για την ε, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα ισχύει μόνο μετά το 2014. Δηλαδή από το 2013 και μετά. Η για την οικονομική διακυβέρνηση αποφασίσαμε ομόφωνα ότι χρειάζεται αλλαγή στη συνθήκη για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά αυτοί οι μηχανισμοί. Ε, όταν τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα ε, πέρυσι, κανεί δεν φαντάστηκε ότι θα προταθούν αλλαγέ τόσο σύντομα. Όμω, όλε αυτέ οι μεταρρυθμίσει δεν είναι ποτέ απλέ διαδικασίε και υπάρχουν πάντοτε ενεχόμενοι κίνδυνοι. Αυτό είναι ένα από του λόγου για του οποίου εξήγησα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και νωρίτερα, ότι δεν θα πρέπει να αποδεχτούμε μια αναθεώρηση τη συνθήκη που να θέσει σε αμφιβολία τα ε, κυρίαρχα δικαιώματα των κρατών μελών. Και βεβαίω αυτή η άποψη έγινε δεκτή. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, οποιαδήποτε αναθεώρηση θα περιοριστεί σε χειρουργική παρέμβαση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πολύ ευθεία και ε, αυστηρή προσέγγιση, προσεκτική. Γι' αυτό συστήνω τη σύνεση και την υπομονή. Θα πρέπει να, να αρχίσουμε να εργαζόμαστε και να μελετούμε αυτό το θέμα μαζί με άλλα θέματα σε σχετιζόμενα. Αξιότιμα μέλη όλες αυτές οι δράσεις δεν ε, είναι κενές νοήματος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Σύνοδος G20, η, ε, το περασμένο Σαββατοκύριακο συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Λισαβόνα, Όλα αυτά είναι μέρο ενό ευρύτερου προγράμματο για να ενισχύσουμε την Ευρώπη και να ξαναέχουμε ανάπτυξη. Στην επόμενη συζήτηση, στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, θα μιλήσουμε για τη σύνοδο του G20. Εδώ ήθελα λοιπόν σύντομα να συζητήσω τα βασικότερα στοιχεία των όσων διεμήθησαν στην ε, συνάντηση Ευρωπαϊκή Ένωση και, Αμερικα... και Ηνωμένων Πολιτειών στη Λισαβόνα το πέρασμα Σαββατοκύριακο. Επικεντρωθήκαμε σε συγκεκριμένα ζητήματα. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο Ομπάμα για την ανάγκη διατλαντικών προτεραιοτήτων και ε, συντονισμού του έργου μα. Για σύγκληση και διαβουλεύσει σε ζητήματα όπω ανταγωνιστικότητα και η παγκόσμια μεταρρύθμιση. Υπάρχουν πολλέ αρμοδιότητε και από τι δύο πλευρέ και ε, το κολέγιο των επιτρόπων θα αναλάβει τι ευθύνε στο πλαίσιο ενό διαπελλοντικού οικονομικού φόρουμ. Και οι αναδυόμενε οικονομίε και το G20 και η παγκόσμια οικονομική κατάσταση απασχόλησε τη συζήτησή μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω θα μπορέσει να πετύχει του στόχου τη μόνον εάν αναλυθεί δράση σε όλου αυτού του πολιτικού τομεί. Αν αξιοποιήσουμε τη σχέση που έχουμε με τι ΗΠΑ σε όλα τα βασικά μα σε, όλες τις βασικές, σε όλους τους βασικούς τομείς. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν την συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο. Ένα πράγμα είναι απόλυτα σίγουρο, ότι θα έχουμε μεγαλύτερη επιρροή αν μπορέσουμε να πετύχουμε συμφωνία μεταξύ μας σε ευρωπαϊκή, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπ' αυτήν την άποψη, ε, ε, με απασχολεί κάπως να απασχολούν πρόσφατε τοποθετήσει κάποιων, οι οποίε δεν συνέβαλαν στο να επικεντρωθούμε και να αποσαφηνίσουμε την κοινή μα προσπάθεια για δράση. Η πρόοδο που έχουμε επιτύχει ω τώρα για την οικονομική διακυβέρνηση είναι ένα δείγμα ότι μπορούμε με επαρκή πολιτική ε, καθοδήγηση από όλες τις πλευρέ να προχωρήσουμε και να προσφέρουμε όφελο σε όλου μα του πολίτε. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό ευρώ, χρειαζόμαστε συνεργασία και σύμπνοια από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ σήμερα. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη συνεργασία και περισσότερο συντονισμό. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων τώρα, ο πρώτος ο πρόεδρος ε, του ΕΛΚ Ζωζεφ Ντόλ. Χθε σε μια δημοσκόπηση, σε μια εφημερίδα διάβασα ότι 70% των Γάλλων λένε ότι η κρίση βρίσκεται μπροστά τους και δεν έχει ακόμα περάσει και λυθεί. Μια ευρύτερη δημοσκόπηση στην Ευρώπη θα έδινε, έδινε τα ίδια αποτελέσματα. Πρέπει να ανταποκριθούμε στα εύλογα αιτήματα των ε, συμπολιτών μας που ανυπομονούν και ενοχλούνται από την καθυστέρηση με την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις. Πολλοί από όσους ε, συνάντησα μου λένε, με ρωτάνε τι κάνει η Ευρώπη, τι κάνει για μένα και την οικογένειά μου. Οι άνθρωποι φοβούνται και βλέπω ότι όλο και περισσότεροι πολιτικοί, όλο και περισσότερες χώρες, ακόμα και σε ή την αίθουσα, χρησιμοποιούν, χειραγωγούν, εκμεταλλεύονται αυτό το φόβο, αυτή την ανησυχία και δεν έχουν να διατυπώσουν προτάσει. Αυτή η λαϊκιστική θέση που επηρεάζει την πολιτική μας είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά και πραγματικά προβλήματα των χωρών μας, της Ευρώπης και του κόσμου. Και νομίζω ότι πρέπει οι πολιτικές ομάδες, οι ομάδες που ε, απορρίπτουν αυτή την λαϊκιστική πολιτική να κάνουν περισσότερα πράγματα δεν μπορεί με τον προστατευτισμό να ληφθεί το πρόβλημα της Ευρώπης. Δεν υπάρχει εύκολη γρήγορη λύση στην κρίση που αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι δυνατόν να γυρίσουμε την πλάτη μας στην αλληλεγγύη σε προσπάθειες που χρειάζονται ώστε η Ευρώπη και όλες οι χώρες μας να γίνουν πιο ισχυρές απέναντι στην παγκοσμιοποίηση αντιλαμβανόμενοι ότι χρειαζόμαστε τους εταίρους μας. Πρέπει να αντλήσουμε ορισμένα διδάγματα από αυτά που συνέβησαν στην Ιρλανδία και Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, πρέπει να λύσουμε λοιπόν διδάγματα από όλες αυτές τις εμπειρίες, διότι τα προβλήματα αυτών των, αυτής της χώρας δεν οφείλονται στις τράπεζες της αλλά και στη δημοσιονομική και πολιτική της κυβέρνησης. Ο κερτικός τίγρης, ο οποίος δημιούργησε την ανάπτυξή του με, τρα, ελάχιστη ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος, με ένα ρυθμό που δεν υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης, αντιμετωπίζει σήμερα την κατάρρευση της στεγαστικής του φούσκας, τεράστια ε, ε, χρέη των ε, νοικοκυριών και ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο έχει στραγγαλιστεί. Πρέπει λοιπόν να λάβουν, θα, θα δοθούν 400 δισεκατομμύρια ευρώ που σημαίνει τρεις φορές το ΑΕΠ του. Θα αντιμετωπίσει λοιπόν τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα. Ζητά λοιπόν δικαιολογημένα σήμερα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και όπως έλεγε ο Υπέτροπος Όλη Ρεν, η βοήθεια που θα δοθεί στην Ιρλανδία θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα όλη τη Ευρωζώνης. Αλλά αυτή η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, την οποία ε, ε, ε, επωφελείται η Ιρλανδική κυβέρνηση, την εφάρμοσε εδώ και χρόνια Πόσες φορές τα κράτη-μέλη προσπάθησαν να προσεγγίσουν, να συγκλίνουν τα δημοσιονομικά του συστήματα ώστε να υπάρχει καλή διακυβέρνηση του ευρώ και κάθε φορά ορισμένες χώρες πάντα οι ίδιες αντιστάθηκαν σε αυτή την προσπάθεια. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να αντλήσουμε διδάγματα από αυτές τις συμπεριφορές για το μέλλον. Το έχω πει κατά επανάληψη σε αυτή την αίθουσα. Μια κρίση είναι ευκαιρία για αλλαγή και δεν πρέπει να φοβηθούμε να αλλάξουμε ορισμένε από τις συνήθειές μας οι οποίες δεν έφεραν τα θετικά αποτελέσματα αποτελέσματα τα οποία περιμέναμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα, μέλα, τα μέτρα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατευθύνσεις που υπέδειξε στη Σεούλ ε, ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να συνεργαστούμε στενά στο πλαίσιο τη Ευρώπη και με, ανάμεσα, και με του μεγάλου διεθνεί συνασπισμού για να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα των χρηματαγορών, να περιορίσουμε τι ανισότητε και να αποφύγουμε μία μάχη, έναν πόλεμο των νομισμάτων. Από μόνε του οι χώρε μα δεν μπορούν να βρουν μία αξιόπιστη και μακροχρόνια απάντηση στα αιτήματα των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Περιμένουν από τους ηγέτες, τους πολιτικούς, από όλους εμάς και από τις πρωτεύουσές μας αποφάσεις που θα καθορίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό που μας δίδαξε η κρίση είναι ότι οι λύσεις σημερινές δεν είναι και οι λύσεις του αύριο πρέπει, θα πληρώσουμε ένα πολύ πιο ακριβό τίμημα αν εξακολουθούμε να αγνοούμε αυτό το πράγμα. Καλό λοιπόν τα θεσμικά όργανα της κυβερνήσης των κρατών μελών μας να αλλάξουν στάση, να αντλήσουν πολιτικά διδάγματα από την κρίση και να μην θεωρούν και να μην θεωρούν ότι χρειάζεται αλληλεγγύη μόνο όταν προκύπτουν προβλήματα. Δεν μιλάμε για διαμάχη μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Μιλάμε για την εφαρμογή της συνθήκης, μιλάμε για την αλληλεγγύη, μιλάμε για συνεργασία. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να σας μεταφέρω, ώστε να μπορέσουμε να, ξεπεράσουμε την κρίση προς όφελος των πολιτών μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επόμενος ομιλητής είναι ο, ο πρόεδρος Μάρτιν Σούλτς, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Ακούγοντας τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διαπιστώνει διαφορετικό ύφος κανείς από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Ρομπέι, αυτά που μας είπατε σημαίνουν ότι όλα ωραία και καλά, μια χαρά τα πάμε. Ακούω τον κύριο Μπαρόζο και διαπιστώνω το εξής. Και παραθέτω, ε, ορισμένες από τις αποθετήσεις που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα δεν οδήγησαν σε περισσότερη συνοχή. Αυτό το λέει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Συμβούλιο, το οποίο μας παρουσιάζεται αγγελικά πλασμένο και ομονών. Όχι. Η πραγματικότητα στην Ευρώπη έχει διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει, διαλύεται σε τρία τμήματα. Γαλλογερμανικό διευθυντήριο, την υπόλοιπη Ευρωζώνη και τις υπόλοιπες χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη με ειδική θέση για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδού η πραγματικότητα στην Ευρώπη. Και ποια είναι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, να την κοιτάξουμε προσεκτικά. Το γαλλογερμανικό διευθυντήριο Μέρκελ ε, Σαρκοζή τα έχει κάνει πλακάκια με τον Κάμερον. Αυτά είναι γνωστά τη πάση, να τα πούμε όμω. Που λέει, εγώ θέλω αναθεώρηση τη συνθήκη για το σύμφωνο σταθερότητα. Οκ, λέει ο Κάμερον. Δεν είναι εύκολο για μένα, γιατί έχω τα ορεινά έδρανα στο ε, κοινοβούλιο μου. Δεν το θέλω να μου δώσετε άλλο προπολογισμό. Και λέει η κυρία Μέρκελ και ο κύριο Σαρκοζή μετά Εντάξει, καλά, ωραία, να το κάνουμε έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ευρώπη. Με κοινοτικό πνεύμα καμία σχέση, αλλά καμία όμως. Αυτή είναι μια διαδικασία που σπάει τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δυνικές θα διαλύσει και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβάμαι ότι ορισμένοι έχουν και συμφέρον και χειροκροτούν ενθουσιοδός απέναντι. Να, συνάδελφοι εδώ κάθονται μεταξύ μας. Όποιος δεν θέλει αυτοί οι άνθρωποι στο μέλλον στην Ευρώπη να έχουν το πάνω χέρι θα πρέπει να φέρει την Ευρώπη σε άλλη κατεύθυνση. Είναι μόνο αυτοί οι τέσσερις εντάξει, λέει η κυρία Χάρμς. Ε, προσπαθώ να συνεχίσω. Ε, ο κύριος Λάγκεν είναι πάντα έτσι ευέξαπτος, το ξέρω. Λοιπόν, η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας έγινε με συμφωνία μια χώρα, μάλλον γίνεται ομοιρία στα χέρια μια χώρα αυτή η υπόθεση που δεν ανήκει καν στο ευρώ. Η κυρία Μέρκελ μιλάει για αναθεώρηση τη συνθήκη σε μια κατάσταση όπου εδώ στο Κοινοβούλιο ουδή δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί στην Ιρλανδία. Εγώ δεν γνωρίζω αν η αναθεώρηση τη συνθήκη στην Ιρλανδία θα περάσει ε, έτσι τόσο εύκολα και τόσο γλυκά όπω μα λέει σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η κυρία Μέρκελ λέει θα πρέπει να συμπεριφθεί και ο ιδιωτικό τομέας. Θέλω να ρωτήσω εσά κύριε Ρεν για τον ιδιωτικό τομέα της Ιρλανδίας. Μα πώς πέρασαν τα τεστ, αυτά τα stress test ε, ε, οι δράπεζες ε, της Ιρλανδίας, το τεστ κοπόσεως. Αυτά που κάνει η κυρία Μέρκελ είναι stress test για το ευρώ το ίδιο. Να σας πω τι γίνεται συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι σωστή, εντάξει, καλή. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιμένω αποφασίσαμε συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με μεγάλη ομοφωνία για ε, ένα φόρο των ε, συναλλαγών και το συζήτησαν λίγο στη Σύνοδο των 8, το απέρριψαν, είπαν όχι δεν θέλουμε φόρο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και το εγκατέλειψαν. Και μετά πήγαν για καφέ. Και το έθαψαν κυριολεκτικά αυτό το θέμα. Θέλουμε να μπει ο ιδιωτικός τομέας, ο συγκεκριμένος ιδιωτικός τομέας, η συμμετοχή του είναι αυτή. Και τώρα μας λένε το Ηνωμένο Βασίλειο δεν το επιθυμεί αυτό. Και δεν κατάλαβα, το Ηνωμένο Βασίλειο κυβερνάει στην Ευρώπη και αποφασίζει για τα πάντα. Και τι γίνεται με την Ευρωζώνη. Στο ιστορικό της Ευρωζώνης, αν εμείς αποφασίσουμε να συμμετέχει ο ιδιωτικό τομέα. Ε, το χρόνο, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Σιγά ηρεμήστε, τελειώνω. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο αγόρευσης. Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Επαναλαμβάνω. Ο κύριος Φαράτζη είπε «Ein Volk, ein Reich, ein Führer» για να το ακούσουν και οι διερμηνείς και να το μεταφράσουν. Ένας λαός, μία αυτοκρατορία, ένας Führer. Mr. President, well, is time is over, please. Έχει τελειώσει ο χρόνο σα, λέει ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Κύριε όλοι ολοκληρώνετε παρακαλώ. Yeah. Yeah. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω αμέσω. Αν αυτός ο συνάδελφος εδώ, αυτός ο κύριος, έρχεται στην αίθουσα και λέει τέτοιες εκφράσεις. Αυτοί που το είπαν στη Γερμανία αυτό το πράγμα, είναι κάποιοι ε, τους οποίους εγώ καταπολεμώ στο πνεύμα τους και στην ιδεολογία τους, αλλά νομίζω πιο κοντά στην ιδεολογία τους βρίσκεται εκείνος παρά εγώ. Ο κύριος Δόλ. δεν μπορώ να δεχθώ αυτό που είπατε βρισκόμαστε σε μια δημοκρατική περίοδο με δημοκρατικά καθεστώτα. απαιτώ να ζητήσετε συγνώμη, να ζητήσετε επίσημα συγνώμη. Αλλιώς, αλλιώς θα σας καταγγείλουμε, θα σας, θα σας μηνύσουμε. Δεν είναι λογικό, δεν είναι δυνατό να λέγονται τέτοια πράγματα μέσα στην αίθουσα. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης για να λυθεί το πρόβλημα. Uh, uh, we must... Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να προχωρήσουμε. Ε, μισό λεπτό. Θα το λάβω υπόψη. Θα το λάβω υπόψη. Θα ληφθεί υπόψη. Μην ανησυχείτε, καταγράφετε. ο πρόεδρος θα ανακαλέσει στην τάξη οποιοδήποτε μέλος που θα διακόψει την ομαλή διεξαγωγή ε, της συνεδρίασης και του οποίου η συμπεριφορά δεν συμμορφώνεται με τον 11ο, με τον του κανόνα 9. Με τον Συνάδελφε, για αυτά που είπε ο κύριος Σούλτς, είναι τελείως αντιδημοκρατικός και φασίστας. Well, uh, uh, uh, we, expected something. Συνάδελφε, κάτι διαφορετικό περιμέναμε, διότι δεν θέλαμε να πάρει τέτοια τροπή η συζήτησή μας. Συνάδελφε, θα πρέπει να συναντηθούμε για να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και να συζητήσουμε μεταξύ μας. Sorry. Sorry. Oh, it is impossible to, to keep... Μπορούμε τώρα να... Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σε αυτές τις συνθήκες, με τέτοια ατμόσφαιρα. Colleague, as you see, the chamber is... Όπως βλέπετε όλοι στην αίθουσα διαμαρτύρονται έντονα κατά τη συμπεριφορά σας. So, it is uh, article number Στο άρθρο 152, σημείο 3, σας διαβάζω το κείμενο. Στη μητρική μου γλώσσα. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση διαταραχθεί επανειλημμένος, ο πρόεδρος μπορεί να στερήσει το δικαίωμα εκφρασής από συγκεκριμένο βουλευτή και αυτό μέχρι το τέλος το πέρας τη συνεδρίαση. Αν το παράπτωμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ο πρόεδρος μπορεί άμεσα να λάβει επιθαρχικά μέσα, χωρίς καν να ανακαλέσει στην τάξη το συγκεκριμένο βουλευτή. Ο γενικός γραμματέας μπορεί στη συνέχεια να αναλάβει να εκτελέσει την εντολή του πρόεδρου ανατρέχοντας τους συνεργάτες του που βρίσκονται παρόντες στην αίθουσα. Συνάδελφοι, όπως βλέπετε, οι περισσότεροι βουλευτές απορρίπτουν πλήρως και διαμαρτύρονται για τη συμπεριφορά σας. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να φύγετε από το ημικύκλιο, παρακαλώ. Συνάδελφοι, όπως ξέρετε, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορείτε να εκφράζετε τις απόψεις, αλλά δεν μπορείτε να προσβάλλετε ένα τον άλλο. Διότι δεν μπορούμε να τηρήσουμε την τάξη στη συζήτησή μας κατά τον τρόπο αυτό. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Γκίφερ Χόφστατ, για τους φιλελεύθερους και δημοκράτες. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι αυτό το συμβάν είναι πάρα πολύ σοβαρό και οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να αντιδράσουν σήμερα να λάβουν κοινή θέση από αυτού και ελπίζω όλες οι πολιτικές ομάδες εκτός από τη δική του να είναι σαφείς και να σας υποστηρίξουν στα μέτρα που ε, λάβατε για να μην επαναληφθεί. Je crois que... Euh, Αυτά που είπε ο κύριος Ντόλ για την Ιρλανδία, διότι μας παρουσίασε μια ολοκληρωμένη ανάλυση για την Ιρλανδία είναι σωστά και θα ήθελα να πω στον Ζωζεφ, αν στην αρχή τη χρηματοοικονομικής κρίσης, Ζωζεφ, είχαμε δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωση για τις τράπεζες τον Οκτώβριο του 2008, όπως είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά απορρίφθηκε από τα κράτη-μέλη, ποτέ δεν θα είχαμε αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ε, αντιμετωπίζουμε σήμερα με την Ιρλανδία. Απορρίφθηκε τον Οκτώβριο του 2008. Είπαν ότι δεν ήταν αναγκαίο. Στη Γερμανία έχουμε αρκετά λεφτά για να λύσουμε μόνοι μας τα προβλήματά μας και είδαμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δεύτερον, ποιο είναι το πρόβλημα ε, τώρα εφόσον η ένταση συνεχίζεται ελπίζω ότι αυτή η σταθερότητα του ευρώ θα επανέλθει αύριο μεθαύριο αλλά πρέπει να δούμε τη σημερινή πραγματικότητα και δεν συμβαίνει αυτό σήμερα γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα αυτά που λέχθησαν χθε από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μαζί με τον κύριο Ρεν στη χθεσινή συζήτηση δεν ήταν πολύ παρόντες στην αίθουσα στη διάρκεια αυτή τη συζήτηση, Αλλά αυτά που είπε ο κύριος Τρισέ είναι πολύ σημαντικά. Είπε ότι το πακέτο δεν αρκεί για να επαναφέρουμε τη σταθερότητα τη Ευρωζώνης. Οπότε έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη ευθύνη εδώ στο Κοινοβούλιο, διότι συναποφασίζουμε για όλους αυτούς τους τομείς. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το δούμε το θέμα σοβαρά. Στην πραγματικότητα, ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο μια, ένα νόμισμα που δεν στηρίζεται από μια κυβέρνηση από μια ενιαία οικονομική πολιτική, από μια ενιαία στρατηγική και από μια μοναδική ενιαία ομολογιακή αγορά. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο. Πιστεύουμε στην Ευρωζώνη ότι μπορούμε να λύσουμε το θέμα με 16 ομολογιακές αγορές, 16 κυβερνήσεις, 16 διαφορετικές οικονομικές πολιτικές. Και αυτό είναι ο ρόλος που καλούμαστε να αναλάβουμε και το συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξουμε είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο μακριά από τι αποφάσει του Συμβουλίου και από τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πρέπει να πούμε ότι ο κύριο Τρισέ έχει δίκιο, διότι εκείνο είναι υπεύθυνο για τη σταθερότητα του ευρώ. Καλούμε λοιπόν το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα να ενισχύσουν το πακέτο, που είναι η μόνη απόφαση που μπορούμε να πάρουμε. Να ενισχύσουμε το πακέτο, να κοινοτικοποιήσουμε και να καταστήσουμε αυτόματε τι Κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Να δημιουργήσουμε μια αγορά ομολόγων στην Ευρώπη. Διότι τα σπρέντ δεν θα εξαφανιστούν μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, μεταξύ Ιρλανδίας και Γερμανίας. Αν δεν υπάρχει ενιαία ομολογιακή αγορά και θα μπορούσε να υπάρξει και μια συμπληρωμα... και θα μπορούσαν να προβλεφθούν οι συμπληρωματικέ αποτελεσματικέ κυρώσει για τι χώρε που δεν τηρούν το σύμφωνο σταθερότητα. Και τέλο, ολοκληρώνω, χρειάζεται μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση που να ενισχύει τι επενδύσει. Και αν η γερμανική κυβέρνηση ε, ζητήσει να αλλάξει το άρθρο 136 τη συνθήκη γι' αυτό, εντάξει, α το κάνουμε αλλά ας κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Και στο άρθρο 136 ας προβλέψουμε μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση για το μάλλον, ουσιαστικές αυτόματες κυρώσεις, ώστε αυτή η αλλαγή της ε, ε συνθήκης που επίκειται να αποτελέσει μια ευκαιρία για το μέλλον της Ευρώπης, μια οικονομική διακυβέρνηση δηλαδή, αυτό είναι που θέλουμε, στην Ευρωζώνη και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Από την ομάδα των Πρασίνων ακολουθεί τώρα. Α, συγγνώμη. Ε, γαλάζια κάρτα. Κύριε Φερχόφστατ, είστε πρόθυμος να απαντήσετε σε ερώτηση. Έχετε γαλάζια κάρτα. Yes, ναι, παρακαλώ. Ο κύριος Ντάρτμουθ, ε, γαλάζια κάρτα. In the event that the commission... Στην περίπτωση που η Επιτροπή πετύχει την οικονομική διακυβέρνηση που ζητά και που εσείς επίσης υποστηρίζετε, τότε πιστεύετε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να λαμβάνει πάντοτε σωστές αποφάσεις. Oh, I think, I Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη την πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά των χωρών που δεν εφαρμόζουν σωστά το, συμφων, το Σύμφωνο σταθερότητα. παρά στο ίδιο το Συμβούλιο, όπου οι ίδιοι άνθρωποι του Συμβουλίου είναι αυτοί που έχουν, ε, εργάζονται για τα κράτη-μέλη και είναι τόσα χρόνια στο Συμβούλιο. Δεν έχω δει καμία χώρα να δείξει με τον δάκτυλο κάποια άλλη χώρα και να λέει δεν εφαρμόζεται το Σύμφωνο σταθερότητα. Τα είδατε το 2004-2005 με τη Γαλλία και τη Γερμανία που δεν εφαρμόζαν το Σύμφωνο σταθερότητα και δεν επευλήθηκε καμία κύρωση κατά καμιά από τι δύο χώρε. Αυτό είναι ο λόγο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, ως ε, ένα υπεύθυνο θεσμικό όργανο με αυτή τη μέθοδο θα πρέπει να ακολουθήσει και να λάβει την ηγεσία στο τομέα αυτό. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάτλενερ, διαδικαστικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, πρόεδρε. Διαδικαστικό. Δεν μπόρεσα προηγουμένως να μιλήσω. όταν διώξατε από την αίθουσα το συνάδελφο του UKIP, αλλά δεν εφαρμόζουμε σωστά τον κανονισμό. Ο κύριος Σούλτς είπε τον Ντάνιελ Φαντεστούπ εδώ μέσα φασίστα και δεν κάνατε τίποτα, ούτε ζήτησε συγγνώμη. Δεν συνέβη τίποτα εις βάρος του κυρίου Σούλτς. Αυτό που κάνει τώρα ο κύριος Σούλτς είναι ακριβώς το ίδιο. Κοιτάξτε, για θέμα, για ζήτημα διεξαγωγή τη συζήτηση τάξη ε, θα πρέπει να απευθυνθείτε αμέσω σε μένα. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε την ε, συζήτησή μα. Κύριε Φάραντ, προσωπική έκκληση. Σα εξέφρασα εγώ τη δική μου άποψη. Σα είπα ποια είναι η δική μου θέση. Και υπ' τη σκοπιά, συνάδελφε, σα ζητώ να μην θέσετε σε εμβολία την απόφασή μου. Επόμενο ομιλητή εκ μέρου των Πρασίνων, η κυρία Ρεμπέκα Χάρμ. Συν Πρόεδρος. Äh, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι σχεδόν δύσκολο πια σε αυτή τη φορτισμένη ατμόσφαιρα να παίρνει κανείς το λόγο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και έκφραση της κατάστασης στην οποία θα μπορούσε να περιέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν γίνει η ευρωπαϊκή πολιτική και πάλι ε, επιμελής και προσεκτική. Εγώ συμφωνώ, όπως και ο Μάρτιν Σούλτς. Ε, η μικρή αλλαγή της συνθήκης που θέλει και χρειάζεται η Γερμανία δεν είναι το πρόβλημα, γιατί η οικονομική κρίση δεν είναι θεομηνία. Το πρόβλημα είναι άλλο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ιδιαίτερα εκπρόσωποι των μεγάλων κρατών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι πλέον σε θέση να φροντίσουν στην παρούσα κρίση να δοθεί κάποια θετική όθηση, μια μικρή σπίθα από τις Βρυξέλλες ε, για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη. Περίεργο είναι, αλόκοτο αυτό. Πόσο γρήγορα αυτό το φιλευρωπαϊκό πνεύμα εξατμίστηκε. Είναι αλόκοτο. Η Γερμανία ως μια χώρα που ήταν τόσο πολύ ε, ε από την αλληλεγγύη και στην παλαιότερη ε, ε, ιστορία της και στην πιο πρόσφατη πώς έχει μπει σε αυτή τη μικροψυχία και τον εγωισμό και δεν μπορεί να βγει η Γερμανία από αυτή την κατάσταση σε μια συζήτηση. Γιατί είναι σωστό τα κράτη-μέλη στην Ευρώπη να ε, έχουν τόσο πολύ συνδέσει τις μοίρες τους. Και κύριε Φαρόμπο, πώς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες που είναι ε, ανασφαλείς, που ανησυχούν, όπως πολύ ωραία είπε ο κύριος Ντόλ. Γιατί δεν μπορούμε πλέον να εξηγήσουμε στην Ευρώπη ε, γιατί θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να προχωρούμε μαζί και έχει να τραβάει ο καθένας τον δρόμο του. Αυτό μας λείπει, αυτή η ομοψυχία και αυτό το πνεύμα και αυτό είναι ένα από τα προβλήματά μας. Επίσης κάτι άλλο που λείπει είναι μια ειλικρινής πολιτική δήλωση Δεν θα σώσουμε τον κάθε Έλληνα ή τον κάθε Ιρλανδό. Τράπεζες σώνουμε από περίπτωση σε περίπτωση. Και η Ιρλανδία δεν είναι μια κατεπίγουσα ε, ανάγκη της Ιρλανδίας, αλλά και της Γερμανίας και της Βρετανίας. Ακόμα και δεν σας αρέσει να τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Αυτή λοιπόν η ειλικρινής δήλωση ε, είναι η βάση της κατανόησης των πολιτών να καταλάβουν οι πολίτε και να συμφωνήσουν με τα όσα αποφασίζονται στι Βρυξέλλες αυτού του κρίσιμου καιρού. Έχει δίκιο ο κύριο Φερχόφστατ, πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Η οικονομική διακυβέρνηση είναι αυτό που θα πρέπει τώρα να λάβει σάρκα και οστά και το γνωρίζουν οι πάντε. Και δεν πάει να μα λέει και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο, ξέρω εγώ, θα αναλάβουν τα απαραίτητα μέτρα με συνέπεια κτλ. Μόλι τα ακούω αυτά αρχίζουν και ανάβουν λαμπάκια και καμπανάκια ακούω γιατί ακριβώς αυτό το φιλοευρωπαϊκό πνεύμα της αλληλεγγύης είναι αυτό που μας λείπει. Θα πρέπει να έχουμε αυτό το βήμα που είναι απαραίτητο και θα ήταν συνεπές για την επόμενη ολοκλήρωση. Εντάξει, μιλάμε για το φορολογικό dumping στην Ιρλανδία και πρέπει να αλλάξει αυτό. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Πότε και πώ θα γίνει αυτό είναι επίση άλλη υπόθεση. Γενικά όμω τα κράτη-μέλη θα πρέπει τη φορολογική του πολιτική να τη συντονίζουν, να συνεννοούνται, αλλιώ θα πάνε πολύ άσχημα τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γίνεται και μια άλλη συζήτηση που δεν θα πρέπει να την κάνουμε πάρα πολύ επιπόλαια γιατί ξεκίνησε από πολύ επίσημα χείλη η συμμετοχή των ε, πιστωτών για την αναδιάρθρωση του χρέους και εκείνων που ευθύνονται άμεσα για την κρίση. Πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω πολύ μεγάλη δυσκολία να κρίνω τι είναι εκεί σωστό και τι λάθος. Γνωρίζουμε ότι έπονται η Ισπανία και η Πορτογαλία και είναι θέμα χρόνου να ζητήσουν και εκείνη την κινητοποίηση του μηχανισμού. θα πρέπει τώρα να συμμετέχουν οι πιστωτές. Είναι καλό αυτό, ε, μας συμφέρει. Ή να πούμε καλύτερα, θέλουμε διακυβέρνηση, οικονομική, μεγαλύτερη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα, φόρο, τέλος ε, στις συναλλαγματικές ε, ε, στις συγγνώμη, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές να πληρώνουν και εκείνοι που βγάζουν λεφτά από αυτές τις ιστορίες αυτό ακόμα δεν το έχουμε αποφασίσει ευχαριστώ πρόεδρος Διακόπτης η κυρία Κέι Σουίνμπερν για τους συντηρητές και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ένα θέμα που έχει απασχολήσει το Συμβούλιο και τη δική μου την εκλογική περιφέρεια τελευταία ε, είναι τελικά η οικονομική κατάσταση στην Ιρλανδία και πώς θα ξεφύγουμε από τα διέξοδα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Εκτιμούμε τις προσπάθειες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά όλοι οι πολίτε στην περιφερειά μου θεωρούν ότι πρέπει να έχουμε και μια σταθερή οικονομική ένωση. Ε, όσα ζητήθηκαν στο Κάρντιφ πρέπει να ακολουθηθούν και θα πρέπει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στι στις, Βρυξέλλε να συζητούν τα θέματα παράλληλα, αλλά λαμβάνουν κοινέ αποφάσει. Πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν την οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό είναι ένα σαφέ συμπέρασμα. Χρειάζονται περισσότεροι κανόνε για την οικονομική διακυβέρνηση και περισσότερη πρόστιμα και Χρειάζεται ανάγκη όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο προπολογισμού να πάψουν τα κράτη μέλη να είναι τόσο εγωιστικά και ο καθένα να σκέφτεται τη δική του τη χώρα. Στο Κάρντιφ, την πρωτεύουσα ε, τη δική μου πρωτεύουσα και σίγουρα και στο Δουβλίνο, ε, όλοι ασχολούνται με το θέμα του πώ δαπανώνται τα κονδύλια. Όλοι πιστεύουν ότι χρειάζεται πρόγραμμα λιτότητα και ξέρουν πόσο χρεωμένε είναι όλε οι χώρε καθημερινά και πόσο χρεώνονται. Ξέρουν ότι πρέπει να ληφθούν σκληρέ αποφάσει. Όμω θέλουν να μπορούν να αποφασίσουν πώ τα χρήματα αυτά θα δαπανώνται το να ζητούμε περισσότερα χρήματα για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, περισσότερη χρηματοδότηση για τον ευρωπαϊκό προλογισμό, όταν πρέπει να περικοπούει ο δημόσιο τομέα τη συντάξη, όταν υπάρχουν διατάξει που του πλήττουν, τότε αυτό για πολλού εκλογεί είναι ένα βήμα προκλητικό. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι δεν έχει κάνει καλή δουλειά στην επιβολή των ίδιων των κανόνων τη και των προδιαγραφών τη εντό τη Ευρωζώνη. Πολλέ φορέ δεν δίνει στου πολίτε κίνητρα για να ε, παράγουν περισσότερο χρήμα. Και αυτό σε στιγμές περικοπής των δημόσιων ε, δαπανών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη-μέλη. Εδώ λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να σεβαστούμε τι ιδιαίτερε πιέσει που δέχεται το καλό μέλο και να ε, έχουμε υπόψη ότι τα επίγοντα σχέδια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα πρέπει να λάβουν υπόψη του ότι θα πρέπει να διαμορφώσουμε ευρωπαϊκό προπολογισμό που να λαμβάνει υπόψη την οικονομική πραγματικότητα τη κάθε χώρα. Ευχαριστώ κύριε μου για την ομιλία σα. Θέλετε απαντήσετε κάποιο ένα ερώτημα για το, τον κύριο Λούκαρτ. E Πιστεύετε ότι τα λεγόμενα ευρωπαϊκά κονδύλια που ανέφερε η ομιλήτρια και που δεν ε, ελήφθησαν όπως έπρεπε από τους εκλογείς, δεν είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιστράφηκαν μόνον εν μέρη και μόνον αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σεβάστηκε τις ίδιες τις υποχρεώσεις της. Τι πιστεύει γι' αυτό η κυρία Μελίτρη. Όπως ξέρει ο κύριος συνάδελφος, Ξέρω πολύ καλά από πού έρχονται τα διάφορα κονδύλια και σέβομαι την πηγή του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Οι εκλογέ όμω θέλουν να υπάρχουν δαπάνε σε ζωτική σημασία προγράμματα και όταν το ΑΕΠ είναι το χαμηλότερο από καμιά άλλη, ε, ε, το χαμηλότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι λοιπόν θα υπερασπίζουμε το δικαίωμα αυτό ελέγχου των συμπολιτών μου καθημερινά. Ευχαριστώ κυρία μου, ο Ο κύριος Μπίσκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν ένα μόνιμο μηχανισμό ε, αλληλεγγύης και διάσωσης για την Ευρωζώνη και το καλωσορίζω πραγματικά, το χειροκροτώ. Επί σειρά μηνών η ομάδα εργασίας Φαν που ε, εργαζόταν και ε, κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα. Αλλά είναι πολύ ανεπαρκή αυτά τα συμπεράσματα έλεγχος ε, στα σχέδια προϋπολογισμού λέτε για να αποφύγουμε μακροπρόθεσμα ελλείμματα. Αλλά ε, βλέπουμε ότι για να βγούμε από την κρίση ε, περιορίζονται πάρα πολλοί δημόσιες δαπάνες. Αυτό δεν είναι μόνο αντιπαραγωγικό, αλλά είναι και αρνητικό. Κανένας δεν φαίνεται να έχει βγάλει τα συμπεράσματά του από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ε, δεν μπορεί μια χώρα που είναι τόσο βαριά χρεωμένη να τιμωρείται με χρηματικά πρόστιμα. Για το σύμφωνο ε, σταθερότητας και ανάπτυξης καταστρέφει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών στην Ευρωζώνη η οικονομία άραγε υπαγορεύει τη δράση της πολιτικής και πάλι ε, θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα της ε, κρίσης. Κοινωνικό ντάμπινγκ, επισφάλεια στην εργασία, περικοπές στην παιδεία. Ε, αυτό θα ε, αυξήσει ε, την επιβάρηση και τις δυσκολίες των κρατών μελών και θα τους δυσκολεύσει και την έξοδο από την κρίση. Δεν έχει νόημα να αυξάνουμε την πίεση σε χώρες όπως είναι η Ιρλανδία, η Ελλάδα ή η Πορτογαλία. Μάλλον θα πρέπει να λυθούν καλύτερα οι μεγάλες ανισορροπίες που έχουμε στον οικονομικό τομέα. Άρα οικονομική διακυβέρνηση. Θέλουμε μια Ευρώπη κοινωνική και δίκαια που να βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης και να κυριαρχεί η πολιτική επί της οικονομίας, να διατηρηθεί αυτό ή αν έχει διαταραχθεί να επανέλθει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Συμπρόεδρος Νάιτζελ Φάρετζ. Καλημέρα κύριε Βαν Ρομπόη. Είστε, έχετε αναλάβει καθήκοντα ε, εδώ και ένα χρόνο. Αρχίζει καταραίει το οικοδόμημα, επικρατεί χάους και ίσως θα πρέπει να γίνετε ο αρχηγός της ομάδας των σκεπτικιστών. Για ρίξτε μια ματιά γύρω σας, δέστε τα πρόσωπα, δέστε το, δέστε το θυμό. Ο, ορισμένοι μοιάζουν, φαίνονται σαν να έχουν δει ένα φάντασμα Προσπαθώντα να διατηρήσουν το όνειρό τους, προσπαθούν να καταργήσουν οποιαδήποτε στοιχεία δημοκρατία από το σύστημα. Και είναι προφανές ότι κανένα από εσά δεν διδάχθηκε τίποτε. Και εσείς, Βαν Ρομπέι, όταν λέτε ότι το ευρώ έφερε σταθερότητα, υποθέτω ότι θα έπρεπε να σας χειροκροτήσω, που έχετε αίσθημα χιούμορ. Αλλά δεν είναι αυτή η νοοτροπία του μπάνκερ ο φανατισμός σας είναι πλέον προφανής. Είπατε ότι είναι ψέμα να πιστεύει κανείς ότι ο έθνος κράτος θα μπορούσε να υπάρξει στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο του 21ου αιώνα. Μπορεί να ισχύει αυτό στην περίπτωση του Βελγίου που δεν έχει κυβέρνηση εδώ και έξι μήνες. Αλλά για όλους τους άλλους εμάς, σε όλα τα κρατη μελη της Ένωσης, κοιτάζουμε τα πράγματα κατάματα και λέμε ότι δεν θέλουμε αυτή τη σημαία, δεν θέλουμε το άνθημα, δεν θέλουμε αυτή την πολιτική τάξη, θέλουν όλα να πάνε στο χρονοδούλαπο της ιστορίας. Σήμερα ε, αντιμετωπίζουμε μια κρίση και τώρα υπάρχει και το θέμα, το πρόβλημα της Ιρλανδίας. Ξέρω ότι η απληστία των Ιρλανδών πολιτικών οφείλεται για αυτή την κατάσταση. Δεν θα έπρεπε να δεχθεί τη φούσκα, τη, τα χαμηλά επιδόγια κτλ. Αλλά, βλέπετε, αλλά δούμε ποια είναι η απάντησή σας. Όταν κατέρε η κυβέρνησή του τους είπατε ότι θα ήταν ανάρμοστο να κάνουν γενικές εκλογές. Ο κύριος Ρεν είπε ότι πρέπει να βάλουν σε τάξη τον προϋπολογισμό τους προτού τους επιτραπεί να ε, ε, προκηρύξουν υπάρξουν γενικές εκλογές. Ποιοι νομίζετε ότι είστε τέλος πάντων. Είστε πάρα πάρα πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι. Η αιμονή σας ε, για τη δημιουργία αυτού του ευρωκράτους σημαίνει ότι είστε διατεθειμένοι να καταργήσετε τη δημοκρατία, να βρεθούν άνεργοι εκατομμύρια άνθρωποι και να είναι φτωχοί, να υποφέρουν ώστε το όνειρό σας για το ευρώ να μπορεί να συνεχιστεί. Αλλά δεν θα γίνει, διότι θα ακολουθήσει η Πορτογαλία με, με, με, με το υπερβολικό του έλλειμμα, είναι η επόμενη στον κατάλογο και μετά θα ακολουθήσει φοβάμαι η Ισπανία και το σχέδιο διάσωσης θα είναι 7 φορές μεγαλύτερο από εκείνο της Ιρλανδίας και μετά δεν θα υπάρχουν πλέον χρήματα και είναι πιο σοβαρό το πρόβλημα πέρα από τα οικονομικά. Αν αφαιρέσουμε τη δημοκρατία και την ταυτότητα των ανθρώπων, το μόνο που τους μένει είναι ο εθνικισμός και η βία. Ελπίζω και εύχομαι ότι το ευρωσχέδιο θα καταστραφεί από τις αγορές προτού συμβούν αυτά που προέβλεψα. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Επόμενος κυρία Αγγέλικα Βέρτμαν. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση χρειάζονται βασικές αλλαγές στην οικονομική πολιτική ε, στην Ευρώπη. Ε, μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία, παρακολούθηση της οικονομικής πολιτικής και καλύτερος συντονισμός για τη διαχείριση της κρίσης. Ε, σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης που θα οδηγήσει σε ευθύνη στην οικονομία για να είναι αποτελεσματικές οι κυρώσεις θα πρέπει εγκαίρως και με βάση την παρακολούθηση ε, των οικονομικών να επιβάλλονται νωρί. Και τέλος ο νέος μηχανισμός διαχείρισης κρίσης σημαίνει ότι μεταξύ άλλων τράπεζες και ασφάλειες μπορούν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή απευθύνω έκκληση να ε, δείξουν περισσότερη αλληλεγγύη επιτέλους απέναντι στους φορολογουμένους. Να πω και κάτι για την Κανκούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μιλήσει εκεί με μια φωνή. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρού είναι ακριβώ ε, ευκαιρία στι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας να επενδύσουμε και να ε, τονώσουμε την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας αυτή. Ακολουθεί τώρα ε, το σύνολο των υπολείπων ομιλητών, η κυρία Μαριάν Τάισεν για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ ε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η κρίση των τραπεζών, η οικονομική κρίση, η κρίση στα δημόσια οικονομικά είναι κάτι που μας ε, δίδαξε στο πρόσφατα παρελθόν και καταλάβαμε πολύ περισσότερο από ότι παλιά τι σημαίνουν κρίσεις. Τώρα έχουμε προβλήματα ε, στην Ευρώπη ε, και αντιστάσεις στο ευρώ και ε, η παρέμβαση και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μας έδειξε ότι η ισχύ και ότι η αλληλεγγύη στην πράξη λειτουργεί. Χρειάζεται όμως να συνεχίσουμε τώρα τις διαρθρωτικές προσαρμογές και να προχωρήσουμε σε μια οικονομική διακυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ας ε, διδαχθούμε από την κρίση αυτή για να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές μας δυνάμεις στο μέλλον. Οι αυστηροί κανόνες και οι απαραίτητοι μηχανισμοί διαχείρισης είναι κάτι που το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ε, για τη διακυβέρνηση και τη μακροοικονομική και τα ελλείμματα και τα χρέη. Οπωσδήποτε για να επανέλθει η εμπιστοσύνη, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη και ε, όλα αυτά να μεταφραστούν σε θέσεις απασχόλησης και ευημερία. Ελπίζω κανείς να μην τρομάξει ε, από τα αυστηρά αυτά μέτρα και τα κράτη-μέλη να μην δακτυλοδείχνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, ένα ε, φόβητρο, σε ένα μπαμπούλα για να το πω έτσι. Χρειάζεται να λάβουμε δράση, αλλιώς η παγκοσμιοποίηση θα μας ξεπεράσει. Διαβάσαμε τα συμπεράσματα κύριε Πρόεδρε και πραγματικά η δική σας ομάδα εργασίας έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά τώρα θα πρέπει να περάσουμε στην πράξη ε, στις προσαρμογές που χρειάζονται και είναι και ευπρόσδεκτες. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, πάνω από το μισό πακέτο της ε, οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να αποφασίζετε με συναπόφαση και ταυτόχρονα ζητάτε fast track. Μα στο ΕΚΟΦΗΝ υπάρχει ε, αρκετό περιθώριο ε, για να διαπραγματεύονται με το Κοινοβούλιο και να διαδραματίζει τον πλήρη ρόλο του το Κοινοβούλιο γιατί αυτό επιθυμεί. Και επίσης το Συμβούλιο δεν θέλει αυτοματισμούς, δεν θέλει να ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου, δεν θέλει αυτόματο μηχανισμό, αλλά θα υπάρξει και ένας μηχανισμός, πρέπει να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός αντιμετώπισης των ε, κρίσεων. Μήπως αυτό θα πρέπει να είναι η επόμενη κίνηση. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω την απάντησή σας. Merci. Our next speaker is... Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χιούς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ένα πράγμα στο οποίο όλοι συμφωνούμε είναι ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είναι πολύ ικανοί άνδρες και γυναίκες. Συναντιούνται κάθε τρίμηνο περίπου και δαπανούν απίστευτα ποσά χρημάτων και χρόνου χωρίς να αποφασίζουν τίποτα. Αποδείχτηκε αυτό από τα πρόσφατα γεγονότα στην Ιρλανδία για τον φόρο των οικονομικών συλλαγών. Συζητήθηκε και, στο Μάιο, και το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο σε κάθε σύνοδο και κάθε συμβούλιο το ανέβαλε για το επόμενο. Και το Δεκέμβριο φαντάζομαι θα ξανασυντηθεί και έπειτα στο Δινικές. Εδώ χρειάζεται να γίνει πραγματικά ένα βήμα στην οικονομική κυβέρνηση με διορατικότητα και αποφασιστικότητα για να έχουμε συντονισμό. Ενώ το μόνο που πετυχαίνουμε ω τώρα είναι η καχυποψία, η αμοιβαία καχυποψία, η έλλειψη εμπιστοσύνη, η αναξιοπιστία και η οικονομική στα... έλλειψη σταθερότητα τελικά αντί για τη σταθερότητα. Είναι σαφέ λοιπόν ότι το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη δεν θα λειτουργήσει, ενώ θα υπάρχει πραγματικό κίνδυνο με το νέο σύστημα που προτείνεται, που θα είναι επιρρεπέ στα κυκλικά προβλήματα και θα θέσει σε κίνδυνο την απασχόληση και τι θέσει εργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να έχει ένα μηχανισμό πιο αποτελεσματικό στην Ευρωζώνη για να μπορέσει να έχει και φορολογική και ε, οικονομική ε, σύγκληση. Όχι μόνο κυρώσει και ποινέ. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα κοινή διαχείριση του χρέου, τουλάχιστον για ένα μέρο των δημοσίων χρεών, τουλάχιστον κατά 60% του ΑΕΠ. Και θα πρέπει τα ωφέλη ενό τέτοιου συστήματο των ευρωπαϊκών ομολόγων να είναι σαφέ και ξεκάθαρο. Κύριε που οι συνεργάτε σα λένε ότι δεν σα αρέσουν ιδιαίτερα οι πολιτικοί που έχουν όραμα. Πιστεύω λοιπόν ότι προτιμάτε την, την τη δράση στην πράξη. Ε, νομίζω ότι τώρα έχουμε αρχίσει να, να φέρνουμε πιο κοντά τα δύο αυτά ρεύματα. Είναι σαφέ ότι αν θέλουμε ισορροπία στην οικονομική διακυβέρνηση, πέραν τη επαγρύπνηση και θέλουμε και κοινή διαχείριση του χρέου, έφτασε πια η στιγμή, πρόεδρε Φαρομπόη, και όραμα να θέσουμε σε δράση και την ίδια τη δράση. Ευχαριστούμε κύριε Χιούς. Ο κύριος Λάνστορφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω κάτι έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουν και οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι χρεωμένη είναι κρίση του χρέους των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω είναι το μόνο πολιτικό επίπεδο στην Ευρώπη που ε, είναι ελεύθερη χρέους και επιθυμώ να παραμείνει έτσι. Αλλά έχουμε ενώσει τις μοίρες μας με το ευρώ και σωστά ε, ε, μίλησε η Ρεμπέκα Χάρμς και ο Μάρτι Σούλτς ε, για ε, έλλειψη εμπιστοσύνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαχειρίζεται τα οικονομικά, όχι οι Υπουργοί Οικονομικών. Ε, και στην Τοβίλ που ήταν πραγματικά μια αποτυχία έπεσε θύμα στην προσπάθεια αυτή ο μηχανισμός. Θα πρέπει να έχουμε οικονομική διακυβέρνηση. Τι είστε η οικονομική διακυβέρνηση που είναι στα στόματα όλων θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπαίνει σε λεπτομέρειες της κοινωνικής πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής, αυτό είναι μεγάλο ερωτηματικό. Ε, θα πρέπει να τονώνονται οι αναπτυξιακές δυνάμεις, εντάξει, αλλά κυρίως τα δημόσια οικονομικά να ξαναμπούν σε τάξη στα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η πρόκληση, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον προπολογισμό και θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ πολύ. Γαλάζια κάρτα. Ο κύριος Σούλτς, ε, Κόμι Λάμστορφ, είστε ε, μέλος του Προεδρείου του Κόμματος των Φιλελευθέρων στη Γερμανία, FDP. Το, αυτό που είπατε τώρα ότι τα ασφάλμα η Ντοβίλ ε, είναι άποψη και του αντικαγγελαρίου της Γερμανίας που είναι πρόεδρος του κόμματός σας ή είναι προσωπική σας άποψη. Είναι θέση του κόμματός σας. Θέλετε να απαντήσετε. Είστε πρόθυμος, βέβαια, είμαι πάντα πρόθυμος να απαντώ. Ο συνάδελφος Μάρτιν Σούλτς είναι και εκείνο στο Προεδρείο της S5 στη Γερμανία και καμιά φορά ε, δηλώνει εδώ πράγματα που δεν συμπίπτουν 100% με τη θέση του κόμματός του. Αν μου δείξετε, κύριε Σούλτς, ποιος ήταν παρόν στην Τοβίλ από πλευράς FTP, ε, θα σας ήμουν ευγνώμων. Και κάναμε και δήλωση σαφή μετά τη συνεδρίαση αυτή. Στην προληπτική φάση ε, ε, ε, εμείς επικρίναμε την κατάληψη του μηχανισμού. Αν γίνει η αλλαγή της συνθήκης θα τα δούμε αυτά, αλλά αυτή η απόφαση της Ντοβίλ ήταν πραγματικά σαφέστατο σφάλμα. Ωραία, ικανοποιήθηκαν οι πάντες από τις εξηγήσεις αυτές, λέει ο Πρόεδρος. Και ακολουθεί ο επόμενος μιλητής ο κύριος Λάμπερτς. Πρόεδρε. Τα κράτη-μέλη έζησαν ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης στηριζόντας την ιδιωτικό χρέος και το δημόσιο χρέος. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το χρέος περιόρισε την κατανάλωση αντί των επενδύσεων, προώθησε την κερδοσκοπία, ενώ η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα είχαν αρχίσει να επενδύουν στα βιβλία ιστορία θα λέγεται ότι ήταν η στιγμή που έχασε σχεδόν τα πάντα η Ευρώπη. Αλλά τίποτε δεν είναι μεραίο. Βεβαίω χρειαζόμαστε στεναρά οικονομική διακυβέρνηση, αλλά αρχικά πρέπει να καταπολεμήσουμε την πυρκαγιά αυτού του χρέου, πιστεύοντα ότι θα λύνουμε το πρόβλημα με τη συμπίεση των δημοσίων δαπανών, σημαίνει ότι αγνοούμε την πραγματικότητα. Δεν θα βγούμε από την κρίση εάν δεν αναδιαρθρώσουμε και δεν ανακατατάξουμε, ανα, ανα, αναδιαπραγματευτούμε το χρέος. Διότι πρέπει να είμαστε σε σαφής Τόσο οι χρεώστε όσο και οι πιστωτέ ευθύνονται για τη συσσόρευση του χρέου. Ορισμένοι δανείστηκαν πέρα από τι δυνατότητέ του, αλλά οι άλλοι παράλληλα δάνειζαν με ανεύθυνο τρόπο, ελπίζοντα ότι θα πετύχαιναν ουσιαστικά κέρδη χωρί κίνδυνο, εφόσον ο φορολογούμενο ήταν πάντα εκεί και να του βγάλει από τη δύσκολη θέση. Και οι μεν και οι δε λοιπόν πρέπει να συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Και αν δεν γίνει αυτό, θα καταδικάσουμε του ίδιου εαυτού μα σε ένα Ιαπωνέζικο σενάριο, σε ένα σενάριο δηλαδή τη παρακμή Ευρωπαϊκή Ένωση, Πιστεύω ότι αξίζουν κάτι το πολύ καλύτερο από αυτό οι πολίτε αυτή τη Υπήρου. Ο επόμενος ομιλητή είναι η κυρία Φόρντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η συζήτηση αυτή αφορά την οικονομική διακυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη. Πολλέ χώρε, και συμπεριλαμβανομένε και τι δική μου, ε, περνούν δύσκολε στιγμέ από οικονομική πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ε, αποστείλει τη βοήθειά του μέσω τη Ιρλανδική θάλασσα. Και δεν είναι αυτή τη στιγμή να αρχίσουμε να καταδεικνύουμε με το δάκτυλο στο Ευρωκοινοβούλιο ούτε χώρε ούτε ανθρώπου, αλλά να λάβουμε καλύτερα αποφάσει για το μέλλον. Ε, την περασμένη εβδομάδα, στα μέσα Νοεμβρίου, η Ελλάδα διόρθωσε για τρίτη αφορά του λογαριασμού τη του τέλου του έτου. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί ένα, ένα πέρα σε αυτή τη διαδικασία. Εάν μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη πρόβλεψη και κατάρτιση των λογαριασμών, θα πρέπει να κλείσει και αυτή η προσπάθεια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει κάνει πολλέ προτάσει για λεπτομερή σχέδια και ανταλλαγή πληροφοριών στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει όλα αυτά να τεθούν επιτέλου σε εφαρμογή. Ναι, βεβαίω πρέπει να ανταλλάσσουμε καλέ πρακτικέ μεταξύ των διαφορών χωρών. Όμω πρέπει επίση να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι όλε οι χώρε στην ίδια θέση. Η καλή οικονομική διακυβέρνηση μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικού τρόπου, προ όφελο όμω όλων. Ευχαριστούμε. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντεμπρίν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν προβλέψει δισεκατομμύρια ευρώ περικοπές στην Ιρλανδία. Θα υπάρξουν ε, σοβαρές μειώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και πολλές δυσκολίες για, αυτούς που έχουν, για τους χαμηλόμιστους. Η ασθενείς, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι θα είναι αυτές οι ευαίσθητες ομάδες που θα πληγούν περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει βοήθεια από την Ευρώπη. Είμαστε τελείως εναντίον μιας τέτοιας βοήθειας. Και αντί να αναζητούμε εντολή για να ε, γίνουν αυτές οι περικοπές τώρα που έβαλαν ε, που μπόρεσαν να βάλουν το πόδι του στη χώρα μα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ε, Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, μα λένε κιόλα να βάλουμε τι εκλογέ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση φαίνεται να μην παίρνει το σωστό δρόμο. Φαίνεται να δρά προ όφελο των φίλων τη τη τράπεζα και όχι του ίδιου του Ιρλανδικού λαού. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μποργκέτσιο. Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Τρισέ, εάν βρισκόταν στη Ρώμη, θα ήταν ένας συγκλητικός με την τίβενό του. Και θα του λέγαμε εμείς τρικέτε πατσιέντσια νόστρα, δηλαδή έλεος κύριε Τρισέ. Είναι σωστό ο δρόμο που παίρνουμε. Πρέπει να υπερασπιστούμε την Ευρωζώνη. Δεν είναι πια δύσκολη επιλογή αυτή. Διότι καταστρέφουμε ουσιαστικά τι οικονομίε των κρατών μελών επιλέγοντα αυτόν τον δρόμο. Η φιλοευρωπαϊκή πολιτική φαίνεται να έχει καταστρέψει τι βιομηχανίε μα και ιδίω τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ιδίω στην Καλαβρία. Σκέφτομαι την ανεργία. Σκέφτομαι το τι συμβαίνει με του συνταξιούχου. Γιατί οι χώρε που επιβιώνουν από την κρίση θα πρέπει να διασώσουν με εκατοντάδε εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ την Ιρλανδία που είχε τόσο χαμηλού εταιρικού φόρου 12,1%. Αθέμητο ανταγωνισμό ήταν αυτό εναντί των υπόλοιπων χωρών. Τι κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μήνα αφού έχει μετά τα τεστ αντοχή ε, και αφού υπάρχει ένα έλλειμμα 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι κάνει ο κύριο Τρικέτ τότε, Τρικέτου στην κλητική. Μα στην Γερμανία υπάρχει και Συμβούλιο Επικρατείας. Συνταγματικό δηλαδή. Και εκεί ε, συζητούνται τα θέματα του ε, γερμανικού ελλείμματος. Τσάω λοιπόν στο ευρώ. όταν έχετε ένα λεπτό να τηρείτε το χρόνο σας. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κύριος Λάγκεν τώρα για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Πολύ κριτική άκουσα για τις αποφάσεις της Ντοβίλ, αλλά οι πάντες γνωρίζουν ότι στην αρχή της περασμένης συνεδρίας της ε, δικής σας ομάδας, κύριε Φαν ε, Task Force, ε, εκκρεμούσαν ακόμα 20 θέματα και επειδή αυτά είναι στην ομοφωνία, κάπου πρέπει να δοθεί μια λύση. Αυτά τα γνωρίζουν οι πάντες, επαναλαμβάνω. Και τα δύο μεγαλύτερα κράτη-μέλη έχουν σφάλει και δεν έχουν τηρήσει το 2004 το Σύμφωνο Σταθερότητας. Και στη Γερμανία κυβερνούσαν οι πράσινοι και οι σοσιαλιστές. Οπότε ο κύριος Σούλτς αυτά που λέει είναι τελείως ε, εκτός τόπου. Ωραία το ε, ε, σύμφωνο σταθερότητας να χαλαρώσει, αλλά θα πρέπει να τα τηρούν τα κράτη-μέλη αυτά που συμφωνούν. Τι να το κάνουμε, να έχουμε οποιαδήποτε σύμφωνα που συμφωνούμε και μετά δεν τηρούμε αυτά που συμφωνούμε. Τώρα έχουμε έξι νομοθετικές προτάσεις. Ε, τα δύο είναι κανονισμοί του Συμβουλίου και δύο είναι κοινοί κανονισμοί Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Δεν καταλαβαίνω γιατί ε, ε, αυτός ο θρήνος εδώ και οι διαμαρτυρίες αφού συμμετέχουμε στη συναπόφαση. Τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγω ρητά θα τις υποστηρίξουμε και μετά να έρθουμε να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Έτσι έχει η πραγματικότητα. Τώρα γιατί εμείς ερχόμαστε εδώ ε, να υβρίζουμε τρίτους που είναι μέλη της νομοθετικής διαδικασίας αντί να κάνουμε τη δουλειά μας. Να πω και δύο λόγια για την αναθεώρηση της συνθήκης. Κατά την άποψή μου η συνθήκη στις 9 Μαΐου ε, έφτασε στα όρια της από το πολύ ξεχύλωμα. Και υπάρχει και το άρθρο 122, αλλά τα κράτη-μέλη δεν το επιθυμούν αυτό, γιατί ε, στη συνέχεια ενδεχομένω να συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι σφάλμα. Και δεν αρκεί να αλλάξει μόνο το άρθρο 136. Χρειαζόμαστε μια νομική βάση για το μηχανισμό ε, διάσωσης, ε, σωστή και γερή και τα υπόλοιπα θα λυθούν. Ευχαριστώ. Η κυρία Φερέρα, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ας είμαστε σαφείς. Ο μηχανισμός, ο μηχανισμός αλληλεγγύης για τις κυρίαρχες οικονομίες δεν έχει λειτουργήσει ούτε θα λειτουργήσει. Δεν διορθώθηκε η ελληνική κρίση. Η Ιρλανδία βρίσκεται σε οικονομική ύφεση. Τίποτα δεν πετύχαμε. Η διαδικασία που ε, δημιουργήθηκε ήταν και καθυστερημένη στη δημιουργία τη και ε, διακυβερνητικά για του ίδιου λόγου που αναλύθηκε και η πρωτοβουλία δημιουργία του ευρώ. Ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα μα προτείνει την ενοποίηση και ενδρέωση του συστήματο αυτού. Όμω, ένα το τρίτο από τα εργαλεία που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν ουσιαστικά μιλά και για ε, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Την πρόταση αυτή την είχαμε ξανακούσει και από την ε, καγκελάριο Μέρκελ και ε, είχαμε καταγγείλει αυτή την πρώιμη ανακοίνωση που είχε διαταράξει τις άγορες. Το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει πλήρως τις ευθύνε του και να ασκήσει πλήρως και τι εξουσίε του σε ένα πνεύμα συνεργασία και στη διαδικασία της συναπόφαση. Ακολουθώντας το νομοθετικό πακέτο για την οικονομική και διακυβέρνηση. Όμω δεν θα πρέπει να θυσιάσει με βιασύνη την ταχύτητα ή την ποιότητα. Ε, ή μάλλον στο όνομα τη ταχύτητα την ποιότητα των ε, νομοθετικών μέτρων. Το Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν θα συμμετέχει ενεργά, αλλά σε ένα τόσο σοβαρό όπω ε, η αντιμετώπιση του δημόσιου χρέου, αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το επιλύσουμε χωρί να λαμβάνουμε υπόψη τα ωφέλη και την προστιθέμενη αξία για του Ευρωπαίου πολίτε. Αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία. Και αυτό που χρειαζόμαστε εμεί ω Ευρωπαίοι είναι ένα σαφέ ευρωπαϊκό όραμα σε αυτήν τη στιγμή, την περίοδο κρίση. Ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αλληλεγγύη και Σταθεροποίηση Αντιμετώπιση του Δημόσιου Χρέου πρέπει να είναι δυναμικό. Πρέπει να παράγει δυναμικά μέσω ευρωπαϊκών συστημάτων και όχι διακρατικών, διακυβερνητικών. Πρέπει να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε με 1% του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Θα πρέπει η αύξηση να ε, μεταφραστεί σε πραγματική σύγκληση, δηλαδή στι πολιτικέ προτεραιότητε τη Ευρώπη. Θα πρέπει ή ο κατάλογο προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή προ... Τη Επιτροπής να είναι κάτι που θα περασπίζεται και ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ένα αποκύημα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Αυτό δεν είναι το πρόσωπο που θέλουμε να δείξουμε στου Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η κρίση της Ευρωζώνης είναι γεγονός και η σοβαρότητα της κατάστασης φαίνεται στα αιτήματα αλλαγή των διατάξεων της συνθήκης της Λισαβόνας που με τόση δυσκολία ψηφίστηκε η Γαλλία και η Γερμανία δεν θέλουν να πληρώσουν για την ελληνική κρίση και την κρίση στις άλλες χώρες. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε το προηγούμενο που συνδέεται με την υιοθέτηση της συνθήκης Λισαβόνας που θα έπρεπε βασικά να διευκολύνει και να απλοποιήσει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ έχει συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Εάν θέλουμε να βάλουμε τάξη, πρέπει να βάλουμε τάξη στο μηχανισμό της Ευρωζώνης αλλά και στους θεσμικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κρίση στην Ελλάδα δεν θα είχε λάβει χώρα, δεν θα είχε επέλθει αν η χώρα είχε διατηρήσει το νομισμά της που θα έπρεπε να εκτιμηθεί με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί περισσότερο η Ευρωζώνη. Ο επόμενος ο κ. Μάουρο, δύο λεπτά. Ε, Πρόεδρε, μία αποτίμηση πολιτικού χαρακτήρα και σε σχέση με όσα υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτηση. Δηλαδή, εμείς ακριβώς τα μέλη των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών οικογενειών κατακρίνουμε τους ευρωσκεπτικιστές γιατί δεν πιστεύουν στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι στην Ευρώπη τελικά δεν πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούμε λοιπόν να καταλογίζουμε στους ευρωσκεπτικιστές κάτι που είναι η δική μας η ίδια ευθύνη. Εμείς είμαστε οι βασικές πολιτικές οικογένειες της Ευρώπης. Και ανέκαθεν είχαμε πολύ μεγάλα φιλευρωπαϊκά ιδανικά και ιδεώδη. Όμω έχει φανεί ότι όλε οι κυβερνήσει που είναι έκφραση των δικών μα ακριβώ πολιτικών οικογενειών καθημερινά φαίνεται να παρακολύουν την ευρωπαϊκή διαδικασία τα μεγά... Ε, ώστε να γίνουν πραγματικότητα τα μεγάλα ευρωπαϊκά οράματα. Είναι πολλέ οι περιπτώσει όπου αυτά που λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τη μέρα τη νύχτα διαλύονται και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε μια επιπλέον ευθύνη. Δεν θα μπορέσουμε να προσανατολίσουμε σωστά την συζήτηση και την ε, υλοποίηση πραγματικά πραγματικών ε, προγραμμάτων. Όπω τα ευρωομόλογα ή την μείωση των εκπομπών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποδείξουμε στου Ευρωπαίους πολίτε ότι είμαστε ακριβώ τα ίδια κόμματα που στι χώρε μα καθημερινά μπορούν να υποστηρίζουν την Ευρώπη και να μπορούν να δείξουν τον δρόμο τη διεξόδου από την κρίση, αναλαμβάνοντα η Ευρώπη και τι δικέ της ε, ευθύνε και τι δαπάνε. Αυτό νομίζω ότι είναι η ουσιαστική μα ευθύνη. Δεν μπορούμε να την ξεχνάμε, διότι ακριβώ η ίδια η φύση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος χάνει και εμεί χάνουμε την αξιοπιστία μα. Και το μόνο που ε, λαμβάνουμε σε αντάλλαγμα είναι άδειε αίθουσε και εκλογέ που χάνουν ε, τον προσανατολισμό του. Το 40% των εκλογών χάνουμε έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει κυρία Ποδηματά. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εάν υπάρχει ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τι αποφάσει του τελευταίου ευρωπαϊκού συμβουλίου αυτό νομίζω ότι είναι ότι δεν κατάφεραν να πείσουν τι αγορέ, δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τι αγορέ. και μια που οι αγορέ τη μέρα μα έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί. Μήπω γιατί πέρα από του αυστηρότερου κανόνε δημοσιονομική ε, πειθαρχία οι αγορέ αντιλαμβάνονται ότι όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουμε αλλά διευρύνουμε το χάσμα οικονομικής και πολιτικής συνοχής εντός της ζώνης του ευρώ; μήπως γιατί ο χειρισμός που επιφύλαξε μια ομάδα κρατών σε μια κατά τα λοιπά σωστή ιδέα όπως είναι η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων ο χειρισμός αυτός φάνηκε να ακυρώνει στην πράξη την προστιθέμενη αξία ενός τέτοιου μηχανισμού στέλνοντας λάθος μήνυμα στις αγορές με κίνδυνο να οδηγηθούμε σε ένα μηχανισμό αυτοεκπληρούμενης προφητείας για την ελεγχόμενη χρεοκοπία και αν επιθυμούμε τόσο πολύ την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα τον επιμερισμό των βαρών γιατί αρνούμαστε πεισματικά να προχωρήσουμε στη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο ευρωπαϊκό επίπεδο και τέλος γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ανάμεσα στην αυστηροποίηση των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας και το μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης κρίσης υπάρχει ένα σημαντικό κενό και αυτό το κενό θα μπορούσε να πληρωθεί εάν αποφασίζαμε επιτέλου να εξετάζουμε σοβαρά τη δημιουργία ενός μηχανισμού κοινή διαχείρισης μέρους του χρέους των κρατών μελών με την έκδοση ευρωομολόγων. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Επόμενο μελήτρια κυρία Χιούμπνερ. μισή λεπτό. Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού στα μεμονωμένα κράτη-μέλη θα διαφέρουν τα επόμενα χρόνια. Το διαφορετικό κόστος για τις ανισότητες θα εξακολουθεί να ισχύει ενώ η οικονομική διακυβέρνηση θα είναι αδύναμη ως διαδικασία ε, ε, εντογενάστε υπό αυτέ τι συνθήκε είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιγόντω να ελέγξει ε, την κατάσταση στα πλαίσια του πρώτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να εστιάσει την προσοχή τη στο scoreboard και στην εφαρμογή του συγκεκριμένα. Ένα σύστημα αυτόματων κυρώσεων θα αλλαγή στη συνθήκη, θα απαιτήσει αλλαγή στη συνθήκη και δεν ξέρω πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε στα πλαίσια της συνθήκης. Γι' αυτό ελπίζω το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν ε, αλλαγές οι οποίες θα καθυστερήσουν τη διαδικασία. Η οικονομική διακυβέρνηση δεν είναι απλό ζήτημα. Επειδή το σύστημα ε, στηρίζεται σε μεμονωμένα κράτη-μέλη που δεν συμπεριφέρονται σωστά η, αυτή η στάση τους μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και στη υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να εξασφαλιστεί η ευρωστία και η οικονομική υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνομαι ότι μία αξιολόγηση επιπτώσεων της οικονομικής οικονομικής διακυβέρνησης θα απαιτήσει χρόνο τον οποίο δεν διαθέτουμε. Τα τελευταία δύο χρόνια η Επιτροπή απέκτησε βαθιά γνώση και κατανόηση της κατάστασης των επιμέρους οικονομιών. Την καλούμε λοιπόν να εξασφαλίσει τη συμβατότητα. Δεν έχετε πλέον χρόνο και μεταξύ εσωτερικών και εσωτερικών ανισοτήτων. Ευχαριστούμε. Να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία από τον ΕΟΧ, τους συναδέλφους από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία, που είναι καθώς και παρατηρητές από την ε, ε, Ελβετική Συνέλευση που βρίσκονται στην αίθουσα. Από την ΕΖΕΣ λοιπόν όλοι οι παρατηρητές που θα συμμετάσχουν στην ε, συνάντηση